προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας. Το λόγο έχει η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά, μετά θα έχουμε ένα catch the eye και κατόπιν ε, τον εξονόμους της τον κύριο Επίτροπο. Ε, η κυρία Τούρουνεν για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εγώ βρίσκομαι εδώ ως πολιτικός και θέλω να κάνω μία έκκληση σε εσά υπό την ιδιότητα της ε, εισηγητρίας. Πολλοί από τους φίλους μου έχουν μείνει άνεργοι τα τελευταία χρόνια. Είναι νέοι με ιδανικά και ενθουσιασμό που αναγκάζονται να περιμένουν στην ουρά να παίρνουν ένα ε, επίδομα ενεργεία να ψάχνουν μια δουλειά η οποία δεν υπάρχει. Εκατομμύρια νέων στην Ευρώπη βρίσκονται σε μια τέτοια θέση. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει με αυτή την έκθεση πρωτοβουλία να προχωρήσει και να ζητήσει να τεθεί το θέμα αυτό και πάλι στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Δεν πρέπει η ανεργία των νέων να καταστρέψει μια ολόκληρη γενιά θα πρέπει νέοι να βρουν μια διέξοδο στην κατάρτιση ή σε νέε θέσει εργασία. Είναι 5 εκατομμύρια τουλάχιστον οι νέοι αυτοί οι οποίοι θίγονται από την ανεργία των νέων, η οποία είναι σε διπλάσια ποσοστά από την ανεργία του γενικού πληθυσμού. Είναι απαραίτητο οι νέοι αυτοί να αντιμετωπίσουν την ανεργία προτού του δημιουργήσει προβλήματα τα οποία θα του συνοδεύουν σε όλη τη ζωή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά η οποία θα γίνει μακροχρόνια άνεργη και επομένω κοινωνικά αποξενωμένη. Αυτό είναι ένα τεράστιο κόστο. Δεν πρόκειται μονάχα σε επίπεδο οικονομικό, πρόκειται για, την, για το κόστο σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν πολύ ψηλέ προσδοκίε από τον εαυτό του και νιώθουν ότι έχουν αποτύχει παταγωδό. Αυτή είναι λοιπόν η δυσκολία ότι η αγορά εργασία αυτή τη στιγμή δεν του παρέχει καμία δυνατότητα. Γι' αυτό εμεί ζητούμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα τα κράτη-μέλη να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση τη ανεργία των νέων και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση των νέων, να αποτελέσει αυτό μια στρατηγική προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσει να υπάρξει μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια καλύτερη κατεύθυνση των νέων κατάρτιση και απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την έκθεση αυτή πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταθέτει συγκεκριμένε προτάσει προ την Κομισιόν και το Συμβούλιο και προσκαλεί και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι κατάλληλε ενέργειε. <clears throat> Ζητάμε καταρχήν να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους, ώστε όλοι οι νέοι κάτω από τα 25 να μην μπορούν να είναι άνεργοι πάνω από τέσσερις μήνες προτού αποκτήσουν και πάλι μια θέση εργασίας ή μια θέση μαθητείας. Δεύτερον, Θέλουμε να υπάρχει μια χάρτα ποιότητος για τους ε, ακαδημαϊκού χαρακτήρα μαθητευόμενους, για τους interns, ώστε αυτή η πρακτική να μην οδηγεί μονάχα σε εκμετάλλευση σε αυτήν η δύναμη εργασία, αλλά να οδηγεί σε πραγματική του κατάρτιση. Είναι επίση απαραίτητο να έχουμε περισσότερε θέσει μαθητείε για του νέου. Και ζητούμε όλα τα κρατημένα να δημιουργήσουν task forces για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της αργίας των νέων και φυσικά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια τέτοια ειδική μονάδα. Τέταρτον, προτείνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μέσα τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τουλάχιστον 10% του Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να δίνεται για σχέδια που αφορούν τους νέους. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η διάκριση κατά των νέων στην αγορά εργασίας, να μην απασχολούνται χωρίς κοινωνικές παροχές. Οι προτάσεις αυτές λοιπόν στον τομέα της ανεργίας των νέων είναι οι δικές μας προτάσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τις κατάλληλες επενδύσεις θα μπορούσε η αγορά εργασίας της Ευρώπης να δώσει περισσότερες θέσεις στους νέους και ένα καλύτερο μέλλον. Θα θέλουμε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μαθητείας για τους νέους. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε ότι μα νοιάζει το μέλλον των νέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Πρώτα η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν 20% του συνόλου λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης οι νέοι αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερες δυσκολίες από τους άλλους όταν προσπαθούν να βρουν μια ικανοποιητική θέση εργασία. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προωθήσουν ενεργά την συμπερίληψη των νέων στην ενεργή ζωή της κοινωνίας. Αυτό όμως δεν γίνεται παρά μόνο εάν υπάρξει ποιοτική παιδεία. οι δυνατότητες των νέων δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς. Αντιμετωπίζοντας τις δημογραφικές αλλαγές θα καταλαβαίναμε ότι οι νέοι μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία και των συστημάτων κοινωνικής περίθαλψης. Τέλος, οι νέοι που ζουν στην Ήπεθρο, σύμφωνα με τις στατιστικές, είναι ακόμη λιγότερο προνομιούχοι από τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία ε, Γετρογιούσκα για ένα λεπτό. η παιδεία για τους νέους είναι μία από τις προτεραιότητες της ίσονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπήρξε πρώτη προτεραιότητα. Πριν από λίγες εβδομάδες καταφέραμε να υπάρξει μια διαπραγματευτική εντολή για τα θέματα αυτά. Η έκθεση της κυρίας Τούρνεν τονίζει ιδιαίτερα πώς θα πρέπει να υπογραμμιστεί και να προωθηθεί η κινητικότητα και η δυνατότητα μαθητείας και απασχόληση για τους νέους. Η έκθεση αυτή είναι ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός και ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο του πόσο σημαντική είναι η παιδεία για τους νέους. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε την κινητικότητα των νέων ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν να πραγματοθεί η στρατηγική Ευρώπη 2020. Θα πρέπει να διευκολύνουμε το να εισέλθουν στην αγορά εργασία οι νέοι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία που είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό θα πρέπει να διαπραγματευτούμε σωστά και να βρούμε τα απαραίτητα χρήματα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Έχω κλείσει τον κατάλογο λοιπόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο ήθελε να λάβει το λόγο. Δεν θα μπορέσει κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανεργία των νέων είναι σοβαρό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε και που έχει επιπτώσεις όλο και περισσότερες στη νεολαία. Στους νέους που μόλις βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και δεν είναι σε θέση να βρουν μία αξιοπρεπή θέση εργασίας το φαινόμενο αυξάνεται σε κλίμακα, σε μέγεθος και μεταφράζεται σε διάφορες αρνητικές συνέπειες στην οικονομία, στο σύνολό της και την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εγγυηθούμε τη σωστή παιδεία και εκπαίδευση των νέων. Πέρα από την εκπαίδευση όμως πρέπει επίσης να εγγυηθούμε και μία σωστή τους πρόσβαση στην αρχή της καριέρας τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τουρόνεν για μια εξαιρετική προσπάθεια. Όπως μας υπενθυμίζουν σκληρά οι στατιστικές της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς εξαιρέσεις, αυτοί που θίγονται κυρίως από την κρίση ήταν αυτοί που είχαν προσωρινή δουλειά, οι γυναίκες και οι μετανάστες. Αυτοί που είχαν προσωρινή δουλειά είναι κυρίως νέοι φυσικά, ήταν κυρίως νέοι και έχουμε τεράστια ποσοστά ανεργία στους νέους τα οποία είχαμε να συναντήσουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από νέους που δεν μπορούν πια να βρουν δουλειά. Η αργή ρυθμή ανάπτυξη η οποία ίσως να επανέλθει σε δύο χρόνια τουλάχιστον, η μεγαλύτερη και χρονικά παρατηνόμενη παρουσία των ε, ηλικιωμένων εργαζομένων, δυστυχώς ε, οδηγούν στη μεγένθηση του συγκεκριμένου προβλήματος. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι είναι πλέον απαραίτητο κάθε χώρας μέλος να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα της ανεργίας των νέων σαν ένα ειδικό πρόβλημα γύρω από το οποίο πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας την οποία πάρα πολύ καλά έκανε η κυρία Τουρούνεν και τη συγχαίρω γι' αυτό ζητά από το συμβούλιο και την επιτροπή μια καλύτερη στρατηγική απασχόλησης και αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο οι νέοι έχουν ανάγκη την ευρώπη αλλά και η ευρώπη έχει ανάγκη τους νέους. η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη είναι όμως πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να λειτουργήσει για ένα πολύ απλό λόγο εάν δεν λειτουργήσει αυτή η σχέση και οι δύο πλευρές θα γίνουν φτωχότερες και οι μεν νέοι έχουν όλη τη ζωή τους μπροστά για να έχουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. η ευρώπη όμως είναι αρκετά γερασμένη για να έχει μια ευκαιρία ακόμη σε τούτους τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Η κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως καταδεικνύει αυτή η έκθεση, η κατάσταση των νέων είναι ιδιαίτερα ζωφερή. Έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες για να βρουν θέση εργασίας. Η ενεργεία των νέων ξεπερνάει κατά μεσόρο το 21% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε ορισμένε χώρες είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και είναι πολύ δύσκολο για τους νέους οι οποίοι έχουν μόλις περατώσει τις σπουδές τους να βρουν μια εργασία με δικαιώματα, με αξιοπρεπή αμοιβή. Αυτό το οποίο μπορούν να έχουν είναι ένα stage, το οποίο πολλές φορές δεν είναι πληρωμένο. Έτσι λοιπόν οι νέοι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη μιας εργασίας με, το, με την οποία μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. είναι μονάχα σε θέσεις μαθητείες οι οποίες είναι κακοπληρωμένες και επισφαλείς. Αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες κατευθύνονται για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή η εκμετάλλευση η οποία δημιουργεί θέση μονάχα χωρίς δικαιώματα. Ευχαριστώ. Κύριος Ρώση για ένα λεπτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να βοηθήσουμε τους νέους. Δεν φτάνει το σχολείο για να εκπαιδεύει τους εργαζομένους του μέλλοντος, αλλά θα πρέπει επίσης και το κράτος να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους. Είναι τεράστια πρόκληση η ανεργία των νέων. Έχουμε βοηθήσει μέχρι τώρα, σαν παράδειγμα, τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των κλιματολογικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να μην τις βοηθήσουμε στην περίπτωση της ανεργίας των νέων. Και δεν θα πρέπει να μένουμε αδιάφοροι στις τρίτες χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων πολύ συχνά νέων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κατάσταση της ε, εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφής. Οι νέοι κάτω από 25 χρονών είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ενεργεία πάνω από 21%. Αυτό είναι το διπλάσιο του μέσου ποσοστού ενεργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, αυτοί οι οποίοι είναι άνεργοι σαν νέοι είναι και στη συνέχεια της ζωής τους πολύ συχνά νέοι. Αυτό οδηγεί σε πάρα πολύ σοβαρές κοινωνικές ε, επιπτώσεις για όλη την κοινωνία μας και για την οικονομική και για την κοινωνική της κατάσταση οι νέοι θα πρέπει να έχουν μια καλή και δίκαια ευκαιρία χάρη σε επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων ώστε να έχουν μια στερεά βάση για περαιτέρω απασχόληση. Ευχαριστώ. Ε, για ένα λεπτό. Οι νέοι μας δεν έχουν προοπτικές. Με την έκθεση της κυρίας Τούρνεν έχουμε την πρώτη κίνηση για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια εξασφαλισμένη, ένα εξασφαλισμένο μέλλον για τους νέους να βγουν από την οικονομική εξάρτηση και να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα μέλλον για τους εαυτούς τους. Εδώ μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Η μαθητεία θα πρέπει να διευκολυνθεί και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι καταχρήστες. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σωστό πλαίσιο ώστε να μην χρησιμοποιούνται οι νέοι σε αυτήν την εργασία αλλά να κάνουν άσκηση μαθητείας υψηλού επίπεδου. Αυτό πρέπει να είναι ένα τμήμα της διαδικασίας κατάρτισης των νέων και όχι η βόλεψη των, εργα... εργοδοτών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προωθήσουμε μια τέτοια χρησιμοποίηση αυτών των ευκαιριών από τους νέους και τις νέες. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε με αφασιστικότητα όλες τις διακρίσεις κατά των νέων. Νέοι χρειάζονται ένα μέλλον και εγγυήσεις για αυτό το μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Λένια, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την έκθεση της κυρίας Τούρνεν. Το θέμα που θίγει είναι πολύπλοκο. Η ανεργία των νέων έχει δύο όψεις. Πρώτον, μπορούμε να, να λάβουμε ορισμένα μέτρα, παραδείγματος χάρη για να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας οι πτυχιούχοι μας. Θα μπορούσαμε επίσης όταν είχαμε μεταρρυθμίσει την ΚΑΠ να το είχαμε θυμηθεί αυτό και να είχαμε προβλέψει κατάλληλα κονδύλια για αυτόν τον σκοπό αλλά και τα υπόλοιπα η άλλη πτυχή είναι το κοινωνικό μας ε, πρότυπο. Πρέπει να εφαρμόσουμε μέτρα ώστε οι νέοι να βρίσκουν θέσεις εργασίας, να μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές τους και να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να εποφελούνται από κοινωνικά μέτρα όπως βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ο κύριος... Ε, έχουμε δύο ακόμα ομιλητές και τέρμα. Uh, ε, Mr. Kelly, one Κύριος Κέλλης, για ένα λεπτό. Η ανεργία των νέων είναι μια τραγωδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τραγικό ότι πάνω από 20% των νέων είναι άνεργοι. Πολλοί από αυτούς έχουν υψηλά προσόντα, πολύ καλή παιδεία και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να έχουν θέσει εργασίες γιατί πληρώνουν τα αμαρτήματα άλλων. Οι χρηματοοικονομικοί τρομοκράτες, οι άπλιστοι κερδοσκόποι τους αφαιρούν την ευκαιρία να ζήσουν και τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να έχουν θέσεις εργασίας. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις μαθητείας για αυτούς, θέσεις εργασίας. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβοπληρωμένες δουλειές, δεν χρειάζεται να είναι golden boys. Μπορούν να είναι απλέ θέσει εργασία θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται, γιατί όσο πιο πολύ μένει κανεί έξω από τον εμφώνα τη εργασία, τόσο λιγότερο μπορεί να προχωρήσει. Αν προωθήσουμε λοιπόν την μαθητεία θα, κάνουμε μια μεγάλη, θα δώσουμε μια μεγάλη υπηρεσία προς τους νέους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Είναι πολύ θετική η έκθεση αυτή. Η ψηφοφορία της εκθέσεως αυτής, ενώ διαπραγματευόμεθα τον προϋπολογισμό για το 2011, είναι ιδιαίτερο εύθετη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την επιθυμία του να καταστήσει την πολιτική για τους νέους κατά προτεραιότητα. Αυτό είναι θετικό, αλλά η πολιτική αυτή δεν θα πρέπει να περιοριστεί στο θέμα της κινητικότητας των νέων. Θα πρέπει να αφορά και τα δικαιώματά τους και περί αυτού πρόκειται. Οι καταχρήσεις που διαπιστώθηκαν στα πλαίσια των στάζ είναι ανησυχητικές και δημιουργούν μια παράλληλη αργορά εργασίας για τους νέους. Αυτοί οι νέοι επαναλαμβάνουν τα στάζ το ένα μετά το άλλο και φύγουν τα δικαιώματά τους έτσι και τα συστήματα φυσικά κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό η τροπολογία μου η οποία θέλει να διασφαλίσει επαρκή επίπεδα ζωής σε αυτούς τους σταζιέρ ήταν ε, κάτι το θετικό. Τελευταίο μιλήτρια η κυρία Νεβεντάλοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω ότι η ανεργία των νέων ξεπερνάει το 20% είναι απαραίτητο να υπάρξει μια επίλυση των προβλημάτων αυτών των νέων. Οι ναι, Νέοι είναι η πιο επισφαλής ομάδα στην αγορά εργασίας. Χωρίς εργασία δεν, μπορούμε να, δεν μπορούν οι νέοι να δημιουργήσουν οι οικογένειες, δεν μπορούν να απεξαρτηθούν από τους γονείς τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξουν απαραίτητε επενδύσει και κίνητρα προ τι επιχειρήσει για να απασχολήσουν του νέου. Όταν βρισκόμαστε σε μια συνολική κρίση, είναι απαραίτητο να μην περικόπτονται οι βοήθειες προς τους νέους. Ο της Επιτροπής, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ κυρία Τούρουνεν, κυρία Συγήτρια καταρχήν, για την εκθεσή σας, η οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και πολύ σημαντική αυτήν την στιγμή πραγματικά που βρισκόμαστε. Όπως τόνισε λοιπόν και μια πλειάδα ομιλητών, η, νεότης, η νεότερη γενιά είναι αυτή η οποία θίγεται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Δεν μπορούμε να κατασπαταλούμε λοιπόν το ταλέντο των νέων μας όταν ο κάθε, ένας στους πέντε κάθε νέος είναι χωρίς, χωρίς ε, καμία προσδοκία απασχόλησης. Η Κομισιόν λοιπόν και εγώ προσωπικά είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον πολύ καλό τίτλο αυτής της έκθεσης για την ΕΣΑΦΕΣ, ότι πρέπει να έχουμε καλύτερε ποιότητα θέσει εργασία για του νέου και είναι απαραίτητο να έχουν την κατάλληλη ε, εμπειρία ως μαθητές και ως τσιράκια σε διάφορες επιχειρήσεις. Γι' αυτό υποστηρίζω την μορφή αυτή απασχόλησης και την σωστή χρήση τους. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις κανονικέ θέσει εργασία όπω υπογραμμίστηκε από πολλού ομιλητές θα πρέπει να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι ο αρνητικό αντίκτυπο τη ενεργεία σε μια ολόκληρη γενιά. Αυτό αντανακλάται και στην πρόταση τη Κομισιόν για τη στρατηγική του 2020. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κατανοήσουμε ότι και οι νέοι θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική και αυτό απαιτεί καλύτερη παιδεία και κατάρτιση ένα μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης των νέων, ένα μεγαλύτερο ποσοστό νέων οι οποίοι έχουν και τα απαραίτητα επαγγελματικά πτυχία και να μειωθεί και το επίπεδο της σχολικής αποτυχίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό η Κομισιόν προβλέπει να έλθει με συγκεκριμένε προτάσει για να αρρωγήσει τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να επιτύχουν του στόχου αυτού. Θα παρουσιάσουμε την πρωτοβουλία Ναυαρχίδο μα το Σεπτέμβριο για την απασχόληση, δίνοντα ιδιαίτερη προστασία, ιδιαίτερη σημασία μάλλον, στις ολοκληρωμένες πολιτικές που συνδυάζουν την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα προωθήσει την απασχόληση με μια πλειάδα πολιτικών, ώστε οι νέοι να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασία. Όλα αυτά μέσα από συγκεκριμένε δράσει, αλλά μπορούν να έχουν μια πρώτη θέση εργασία οι νέοι και να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα στην αγορά εργασίας. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο μέτρα υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών και να αυξήσουμε τις δυνατότητες απασχόλησης των νέων, επίσης στοχευμένες δράσεις για τους νέους οι οποίοι έχουν χαμηλά προσόντα και δεν έχουν δυνατότητα να μπουν στην αγορά εργασίας. Συμφωνώ λοιπόν με τους ομιλητές πρέπει να αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένα μέτρα την ανεργία των νέων, να σταματήσουμε αυτή την κατασπατάληση τη ενεργητικότητα και των ταλέντων των νέων ανθρώπων στην Ευρώπη και είμαι σίγουρο ότι με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρούμε το σωστό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε. <clears throat> Λίγη συζήτηση αυτή τη έκθεση. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση τη κυρία Γκρουνή άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου.